Good afternoon, colleagues. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Αν μπορούμε, μπορούμε να, αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρία. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Το πρώτο σημείο στη μέση διάταξη είναι η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για την μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών μας με την θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή. Κύριε Μωράης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, χρειαζόμουν λίγο νεράκι. Ευχαριστώ, Κίνγκα και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την παρουσία τους. Ξέρω ότι είναι πέμπτη απόγευμα και αυτή είναι μια παρουσίαση της ε, έκθεσης αυτής που είναι σημαντική. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα διαβάσουν την έκθεση και άλλοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που βοήθησαν τη δημιουργία αυτής της ε, έκθεσης με τη βοήθεια των εγγράφων εργασίας των συναδέλφων που με βοήθησαν να δημιουργήσω την κύρια έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων για τη μαζική παρακολούθηση. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση. Κράτησε περίπου έξι μήνες αυτό το εγχείρημα. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες από τον κύριο Σνόντεν αλλά και στο ίδιο αυτό πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξαν ρόλο και οι δικές μας εξελίξεις ιδίως για, για τον κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων και πιστεύω ότι και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε Καλή σημαντική επεξεργασία των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Μέσα στους έξι μήνες λοιπόν έγιναν όλες αυτές οι προσπάθειες και ευχαριστώ και τη γραμματεία μας η οποία εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να καλέσει μια σειρά από μάρτυρες και εμπειρογνώμονες που μας βοήθησαν να συντάξουμε αυτή την έκθεση μαζί με τα σημαντικά έγγραφα εργασίας και να καταλήξουμε σε αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο σας παρουσιάζω σήμερα. Το έγγραφο αυτό εργασίας βασίζεται σε τρία στοιχεία ή μάλλον δίνει τρία βασικά συμπεράσματα. Έχουμε καταρχήν τα βασικά ευρήματα και μετά μία σειρά από συστάσεις. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά γιατί είχαμε πολλούς μάρτυρες στις έρευνές μας. Ακούσαμε τις απόψεις πολλών ειδικών από καταγγέλλοντες, σε δημοσιογράφους, επιτροπές που, μέχρι επιτροπές που κάνουν κοινοβουλευτικού χαρακτήρα εποπτεία, μέχρι τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Φυσικά δεν είμαστε ιατροδικαστές, δεν είμαστε δικαστές, απλώς συλλέξαμε πρωτογενείς και δευτερογενείς πληροφορίες που είναι κυρίως περιστασιακά στοιχεία βάσει των οποίων προσπαθήσαμε να συμπληρώσουμε το παζλ. Όπως θα έκανε και οποιοδήποτε εθνικό σώμα και εμείς ως ερευνητικό σώμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να δούμε τη συνολική εικόνα σε σχέση με τις καταγγελίες του Έντουαρτ Snowden και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Επίσης ε, μας είχαν επιφορτήσει στα πλαίσια αυτής της έρευνας με τη διατύπωση μιας σειράς συστάσεων για το μέλλον σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, σε σχέση με τον τρόπο συλλογής δεδομένων με στοιχεία πολιτών και της μαζικής παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίναμε την κατάσταση στις ΗΠΑ με την κατάσταση στην Ευρώπη και είδαμε και τα θέματα του μέλλοντος, πώς πρέπει να λειτουργήσει η προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον έναντι των ΗΠΑ. Έχουμε λοιπόν αυτά τα 18 πορίσματα στην έκθεσή μας που βασίζονται στα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε από την έρευνα αυτή, από τις διάφορες πηγές που προανέφερα κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. Οι συστάσεις και το σχέδιο προτεραιοτήτων βασίζονται σε αυτά τα ευρήματα, τα πορίσματα. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των συστάσεων, οι συστάσεις αυτές βασίζονται και στην εμπειρογνωμοσύνη πολλών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μονάχα στα στοιχεία που μας έδωσαν οι εμπειρογνώμονες που θελήσανε να τονίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ακόμα και πριν ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Το θέμα του SWIFT, του Safe Harbor, του PNR, όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας είναι πια ιδιαίτερα οικεία ήταν ζητήματα που οι κοινοβουλευτικοί της Επιτροπής μας ήδη τα επεξεργαζόταν πριν ξεκινήσει αυτή η κοινοβουλευτική έρευνα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει οριμάσει μετά από πολύ χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να προχωρήσουμε γιατί με τον τρόπο αυτό κατά τη δική μου άποψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεπερνάει την προσέγγιση που είχαν τα Εθνικά Κοινοβούλια αυτό το θέμα. Εμεί θα πρέπει να το ατενίσουμε το ζήτημα αυτό ως αρμόδιοι για πάρα πολλά θέματα προστασία προσωπικών δεδομένων, γιατί ήδη έχουμε επεξεργαστεί τα θέματα αυτά σε νομοθετικό επίπεδο και το κύριο θέμα το οποίο μας απασχολεί σε σχέση με την έκθεση Albrecht για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον κανονισμό και την οδηγία, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά από χρονική έποψη, γιατί μας απασχόλησε αυτό το σημαντικό τμήμα <clears throat> νομοθετικής ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή που συνεχιζόταν η έρευνα μας. Ελπίζω λοιπόν θα έχετε τον καιρό να κοιτάξετε αυτό το έγγραφο εργασίας, το σχέδιο εκθέσεως και τα 18 συμπεράσματα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που εξέτασαν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι παρόντες και αυτοί ακόμα που δεν είναι παρόντες θα ήταν σκόπιμο να δουν τα συμπεράσματα και το σχέδιο προτεραιότητος και όταν το πράξουν αυτό δεν θα πρέπει να το δουν όπως θα το έκανε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά με την πεποίθηση ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε οι αρμόδιοι για να, να βρούμε κάποια λύση για τα θέματα αυτά προστασίας προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσω τα επόμενα σχόλιά μου στις ε, συστάσεις μας, γιατί εκεί είναι που η έρευνά μας έχει τη μεγαλύτερη σημασία και βασίζεται και στα έγγραφα εργασίας των συναδέλφων. Περνάω λοιπόν σε αυτές τις ε, συστάσεις και αναφέρομαι και στα οικία έγγραφα πρώτα απ' όλα για τις συστάσεις αυτές. που είναι και τα στοιχεία από τον οποίων βασίστηκε η διατύπωση αυτής της έκθεσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε πώς πρέπει να διαρθρωθεί το μέλλον της προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο θα έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό χάμπεας κόρπους, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Και επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του λεγόμενου ασφαλούς λιμένα, safe harbor. Εδώ το έγγραφο του κυρίου Βος είχε ζητήσει από την Κομισιόν να αναστείλει την αρχή αυτή του safe harbor που επιτρέπει τη μεταφορά στις ΗΠΑ στοιχείων των ευρωπαϊκών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνθήκη TFTP βάση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, ζητούμε την αναστολή της τωρινής συμφωνίας TFTP μέχρι ότου οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ψήφισμα έχουν εκπληρωθεί. Η Επίτροπος Μάλστρομ ε, κατέληξε μετά από μια διαδικασία διαβούλευση με τι ΗΠΑ ότι δεν υπήρξε παραβίαση τη συμφωνία TFTP. Αλλά αυτό βασίζεται μόνο στι διαβεβαιώσει που μα έδωσαν οι ΗΠΑ. Εμεί θα θέλαμε να συνεχίσει η ενδελεχή έρευνα μαζί με του εταίρου μα των ΗΠΑ για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Θέλω επίση να σα υπενθυμίσω ότι η συναδελφή μου Σοφίν Τβέλτ και η Κορνιλία Έρνστ έκαναν σημαντική εργασία στα έγγραφα εργασία σε σχέση με την με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μηχανισμούς εποπτείας. Είναι κέρια σημαντικό στην έκθεση αυτή να δούμε πόσο σημαντική και ποια είναι η αξία αυτών των μηχανισμών εποπτείας και πώς μπορούμε να ζυγίσουμε τις ε, σχέσεις που υπάρχουν μέσα στις διάφορες υπηρεσίες στο φως των αποκαλύψεων που έγιναν και επίσης πώς μπορούμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη όπως είπα προηγουμένως για την ε, προστασία δεδομένων, η εκθεσή μας ζητά από το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως την επεξεργασία του πακέτου για την προστασία δεδομένων, ώστε να μπορέσει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν και τονίζει επίση και τη σημασία και τη οδηγία και του κανονισμού για, τα, για την προστασία δεδομένων ότι πρέπει να εγκριθούν από κοινού ω πακέτο. του Κοινοβούλιο έχει ήδη δώσει ένα στεναρό μήνυμα και ο εισηγητή ε, κ. Άλμπερτ είναι έτοιμο να συνεχίσει την επεξεργασία η συμφωνία με τις ΗΠΑ στην προστασία των δεδομένων, η συμφωνία ομπρέλα όπως αναφέρεται, είναι κέριου χαρακτήρα και ζητούμε από την Κομισιόν μέχρι την άνοιξη του 2014 να τελειώσει την επεξεργασία και να εξασφαλίσει την έγκρισή της. Ο στόχος είναι να υπάρξει η νομική δικαστική μαλλοθεραπεία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εκτεθεί τα στοιχεία τους μετά από αίτηση των ΗΠΑ και το βασικό στοιχείο που έχει να κάνει με τη μαζική παρακολούθηση είναι ότι ο στόχο μα είναι να εξασφαλίσουμε την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν έχουν μία αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την δικαστική θεραπεία στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών που εγγυάται μονάχα το, η νομοθεσία στους Αμερικάνους πολίτες, είναι δύσκολο να υπάρξει εμπιστοσύνη σε σχέση με τις μεταφορές δεδομένων. Για την TFTP επίσης η έκθεση, την TIP μάλλον, η έκθεση αναγνωρίζει το σημαντικό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι για την οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης πρέπει να εξασφαλίσουμε στεναρές ε, ρήτρε προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων για προφανείς ε, λόγους. Επίσης για την, το υπολογιστικό νέφος αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υπάρξει προστασία για τα δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται αποθηκευμένα στον έφος, γιατί ό,τι βρίσκεται στον έφος μπορεί δυνητικά να τύχει πρόσβαση από την NSA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απαραίτητο επίση οι επιχειρήσει να εφαρμόσουν υψηλού επίπεδου κανόνε για την προστασία δεδομένων και όταν η αποκάλυψη αυτών των γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε, σε απώλεια εμπορικών συμφερόντων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης η Επιτροπή μας άκουσε πολλές απόψεις από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφους για τους καταγγέλλοντες και την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία και πιο εύρωστη προστασία των καταγγελόντων στον πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα της συλλογή πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες. Και ακούσαμε και από δημοσιογράφους όπως από άλλες Ράσπερτ από τον Guardian που αντιμετωπίσανε ε, προβλήματα σχεδόν ανατριχιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την αποκάλυψη των ε, στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σνόουντεν μέσω αυτών. Σε όλη αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια προστασία για τις αποκαλύψεις σε σχέση με τις ε, ε, τεχνολογίες πληροφοριών. Αποκαλύφθηκε μια σειρά από αδιαναμίες του πλαισίου πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παρέμβαση hackers πριν από μερικές εβδομάδες που μπορέσανε να παρισφρήσουν και να έρθουν σε πρόσβαση προσωπικών δεδομένων ευρωβουλευτών χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι παραμένει ένα πρόβλημα ασφάλεια στα ευρωπαϊκά ιδρύματα σε σχέση με την πληροφορική και όπως είπα προηγουμένως πρέπει να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής και έχουμε εδώ μια σειρά από παραγράφους που έχουν προσφέρει οι συναδελφοί μας από άλλες επιτροπές και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και υπάρχουν και πολλές συζητήσεις που κάναμε με τους ομολόγους μας στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι σαφές ότι δεν είναι θέμα διπλωματικών σχέσεων μονάχα, αλλά πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του γεγονότος ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτέ τι επαφέ, οι οποίε θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένε δράσει. Και η πρόσφατη διαδικασία αναθεώρησης που εκκίνησε ο Λευκό Οίκο και η συνέχιση της παρακολούθησης των δικαστικών ε, ενεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Τέλος, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι, προσπαθώ να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πω, συναδελφοί, ότι το κείμενο της έκθεσης αυτής θέλει να ρίχνει ένα διορατικό βλέμμα προς το μέλλον και να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι συστάσεις δεν θα εξατμιστούν μόλις λήξει αυτή η θητεία, αλλά θα έχουν και μια πρακτική συνέχεια. Θέλουμε η στήριξη να εξακολουθήσει και στην επόμενη θητεία και να υπάρχει ένα αποτύπωμα που να χρησιμοποιήσουν τα θεσμικά όργανα στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό καλό τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus και να γίνει θεματοφύλακα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θεσμικά της όργανα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτό που ξεκινήσαμε να προτείνουμε το 2013, ώστε όλε οι συστάσει που κάναμε στην έκθεση κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν. Μην μείνει ένα στατικό κείμενο, ένα καινογράμμα που θα μπει στο ράφι η έκθεση αυτή, αλλά να έχει και πρακτική εφαρμογή. Θέλουμε λοιπόν από το έγγραφο αυτό να ξεκινήσει ε, η πορεία προς την επόμενη θητεία. ώστε να αντιλήσουμε από τι ειδικέ γνώσει περιοδικού βίου που συγκεντρώσαμε και συλλέξαμε σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου μέχρι την επόμενη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτή την ε, συνοπτική παρουσίαση. Να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, αλλά θα πρέπει να ζητήσω και την ε, κατανόησή σας, διότι ο κύριος Σαλαφράγκα της Επιτροπής ΑΘΕΤ πρέπει να φύγει. Οπότε αν δεν σας πειράζει θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο από την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό και μετά θα περάσουμε στον κανονικό κατάλογο αγορητών και τους κοιόδης εισηγητές δηλαδή. Ευχαριστούμε. Κυρία Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές γιατί πράγματι έχω μια πτήση στις 3. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μωράης γιατί είχαμε εξωτερική συνεργασία. Είδαμε ότι υπάρχουν 16 παράγραφοι στο σχέδιο έκθεσής του που αφορούν ε, πιο πολύ την εξωτερική πολιτική και περιορίστηκε πιστά, θα έλεγα, ε, στους όρους του εγγράφου εργασίας ε, που με τους δύο συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε υποβάλει. Βέβαια, υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν βελτίωσης 50 αιτιολογικές σχέσει 116 παράγραφοι συνολικά. Φιλόδοξο το εγχείρημα, είναι και το θέμα άλλωστε πολύ σημαντικό, οπότε μπορούμε να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές της έκθεσης. Μία από αυτές είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη σημασία που έχει η συνεργασία για την καταπολέμηση της δημοκρατίας ε, ε, ε, και με τις ΗΠΑ ένθεκα κίνδυνο, δηλαδή και, από, και για εδώ και για τη ΣΥΠΑ. Τώρα να πω ε, γρήγορα γρήγορα για τις συγκεκριμένε παραγράφους κάποια πράγματα. Θα ήθελα στην παράγραφο 6 θα μπορούσαμε να την να ε, εντάξουμε, ε, ε, εστιάσουμε περισσότερες πρακτικές συνέπειες στην παράγραφο 19 που μιλάει για condemnation in the strongest possible terms, καταδίκη, πλέον περίφραστη καταδίκη Φυσικά και είναι απαράδεκτες τέτοιες δραστηριότητες, αλλά στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι διατυπώσατες που τις χρησιμοποιούμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή μαζικά εγκλήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σεβαστούμε το πνεύμα, ε, διαλέγοντα μια άλλη διατύπωση, είναι συνεπή γιατί θέλουμε σίγουρα στου αυτούς τους παραλογισμούς να τους τονίσουμε, αλλά μέσα στα ωραία. Στην παράγραφο 59 που είναι ιδιαίτερα ευαισθητή και με άλλους συναδέλφους ε, στα μέλη ε, και της Βουλής Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των Ηνωμένων ε, Πολιτειών στείλαμε κάποια έγγραφα λέγοντας ότι μετά από όλα αυτά θα είναι δύσκολο εμείς να υπογράψουμε τη συνθήκη εμπορίου και επενδύσεων είναι ένα θέμα λεπτό, αλλά επειδή είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, πρέπει να βρούμε και την κατάλληλη διατύπωση στο κείμενο. Να είμαστε λίγο πιο λογικοί σε αυτά που λέμε. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω εδώ ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά κυρία Πρόεδρε τον εισηγητή για τη συνεργασία του, το ανοιχτό του πνεύμα. Και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία που είχαμε και ε, με την Επιτροπή αυτή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεχιστεί και σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας, δηλαδή κατάθεση τροπολογιών, εξέταση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράνκα Να περάσουμε στους κοιότητες εξηγητές. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα πολύ καλό υπόβαθρο, είναι μια πολύ καλή βάση για την περαιτέρω επεξεργασία. Εμείς πρέπει να έχουμε την κατάλληλη εποπτεία, να έχουμε τα αιτήματα τα οποία αρμόζουν σε ένα κοινοβούλιο όπως το δικό μας, καλύπτει πάρα πολλά θέματα και αντιμετωπίζει από πολλές οπτικές γωνίες τα θέματα αυτά τα οποία έχουν αναδειθεί στην επικαιρότητα και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ σωστό έδαφος για να μπορέσουμε να προβούμε σε μια αξιολόγηση της συνολικής αυτής δραστηριότητας μαζικής παρακολούθηση. Αν δούμε ποιοι είναι οι στόχοι με τους οποίους εμείς ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, ήταν καταρχήν να επαναφέρουμε το, την εμπιστοσύνη για τις μελλοντικές επικοινωνίες. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη, αλλά και διατλαντική φιλία. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανακτήσουμε και πάλι τον έλεγχο των δικών μας προσωπικών στοιχείων και να κάνουμε πιο ασφαλείς τις επικοινωνίες μεταξύ Ευρώπης και άλλων τμήματων του κόσμου. Να προστατεύσουμε τα ιδιωτικά δεδομένα των ε, πολιτών αλλά και των εταιριών, αλλά και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις όλων αυτών των δεδομένων και φυσικά και σε τελική ανάλυση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προστατεύσουμε καλύτερα από την παρακολούθηση και τις κυβερνοεπιθέσεις. Για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε να υπάρξει μια ρύθμιση σε, δια, σε διεθνές επίπεδο, αυτή η λεγόμενη συμφωνία κατά της κατασκοπίας όπως αναφέρεται. Πιστεύω όμως ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτή η συνολική συμφωνία, συμφωνία ομπρέλα είναι απαραίτητη όπως αναφέρεται και στην έκθεση και είναι απαραίτητο ο μηχανισμός Safe Harbor ο οποίος ε, έχει δημιουργήσει πολλά μειονεκτήματα για τους πολίτες, θα πρέπει να τροποποιηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμοστεί στις τεχνικές μεταλλαγές που λαμβάνουν χώρο, χώρα και φυσικά πρέπει να ανασταλεί μέχρι τότε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα εμπορικής κατασκοπίας και θα πρέπει να εστιάσουμε και περισσότερο στο πώς μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο οργάνωσης των μυστικών υπηρεσιών, ώστε από τη μία πλευρά να μπορούν να εξασφαλίσουν την άμυνα και την προστασία των κρατών μελών και των θεσμών και των ευρωπαϊκών, από την άλλη πλευρά όμως να μπορέσει να δημιουργηθεί μια βάση ώστε να εξασφαλίσουμε ένα κοινό πλαίσιο προστασίας με τους εταίρους μας και με τρίτες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα και γι' αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία <clears throat> κίνηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερες τεχνολογικές ικανότητες και εδώ αναφέρθηκε η τεχνολογία της, του υπολογιστικού νέφους. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε και η διαδρομή των στοιχείων στο ίντερνετ και η κρυπτογράφηση η οποία χρησιμοποιείται για τα πακέτα του ίντερνετ να γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελέγξιμα από την Ευρωπόλ και το κυβερνό κέντρο της Europol γιατί έχω την εντύπωση ότι η Europol μέχρι στιγμής δεν έχει και οι ΕΝΙΣΑ δεν έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα βασικά στοιχεία πρέπει η ενίσα να προχωρήσει για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες αυτές με τις οποίες θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη προμήθεια και λογισμικού στην Ευρώπη, ώστε να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και να σκεφτούμε και καλύτερα για τις προμήθειες που γίνονται σε ευαίσθητους τομείς, αν μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο διενέργειας αυτών των διαγωνισμών. Αυτές θα ήταν οι προτάσεις μου και επειδή και εγώ πρέπει να φύγω, δυστυχώς δεν θα ακούσω τις απαντήσεις του εισηγητή, αλλά γενικά θέλω να επενέσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για το έργο του. Ευχαριστούμε κυρία Ίνφελτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές για το έγγραφο που έχουν ετοιμάσει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό ε, ε, έγγραφο με την έννοια ότι καλύπτει πάρα πολλά θέματα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που είμαι μέλος αυτού του κοινοβουλίου. Φαίνεται να είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο που κάνουμε αυτού του είδους το έργο στην Ευρώπη. Ε, και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατά πρώτον, να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή. Αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να εγκριθούν συνολικά σαν ε, μια δέσμη συστάσεων που θα αφήσουμε ως ε, κληρονομιά στο επόμενο, στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου για να αναλάβει την υλοποίησή τους. Σε αφορά την προστασία, καλά λέτε ότι εδώ και πολλά χρόνια το εξετάζουμε το θέμα αυτό. Είναι μια από τι προτεραιότητε και δεν είναι τίποτε το καινούριο, αλλά γίνεται όλο ένα και πιο επίγον. Τώρα που το πακέτο αυτό εγκρίθηκε και άρα τα πρότυπα που έχει θέσει το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Βέβαια βρίσκω ανησυχητικό και αρκετά ε, δυσάρεστο που τα κράτη-μέλη πέρα από όλε αυτέ τι αποκαλύψει προσπαθούν να αποδυναμώσουν ε, τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων. Καλωσορίζω τις συστάσεις για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών, διότι αυτό το συζητούσαμε ήδη όταν ε, ετοιμάζαμε το έγγραφο εργασία. Επίσης, σημαντικό είναι να δούμε το θέμα της επιβολής, της ισχύω για το θέμα. Δεν είναι απλώς να προβλέπετε νέα νομοθεσία ε, Λόγω χάρη έχουμε καλή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ήδη σε ισχύ. Όμως, ακόμη και αν χρειάζεται μια σχετική επικαιροποίηση, ένα φρεσκάρισμα, υπάρχει. Υπάρχει και ήδη έχουν παραβιαστεί τους ή άλλους οι υπάρχοντες νόμοι. Γι' αυτό λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηροί ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας, διότι εάν πάλι εγκρίνουμε μια τελείως καινούργια νομοθεσία, αλλά δεν παρακολουθούμε το πώς επιβάλλεται, το πώς εφαρμόζεται, τι νόημα έχει. Δεν μπορεί όλα να παρακάμπτονται από τους νόμους μιας τρίτης χώρας, της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Τότε γιατί να καθόμαστε να περνάμε νομοθεσία. Έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε. υπ' αυτήν την έννοια, η μία έρευνα από τα κάτι μέλη και τη Europol για τις εικασίες παραβίασης του συστήματος SWIFT στις κάτω χώρες είναι κάτι που καλώς σημειώθηκε από την ομάδα εργασίας 29. Ε, Νομίζω οι Ολλανδικές και Βελγικές αρχές ε, διεξάγουν μια κοινή έρευνα διεξαγάγουν μάλλον μια κοινή έρευνα, οπότε θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις τους και να προσπαθήσουμε αυτά τα συμπεράσματα να τα καλύψουμε στο κείμενο. Να θυμίσω επίσης τους συναδέλφους ότι αυτό το σώμα, εγκρίνοντα την έκθεσή μου προδιετία, ε, ζήτησε την εκβάθρον αξιολόγηση της ε, σχετική πολιτική μα. Αυτό θα ήταν καλό να το ξαναδούμε από το φω των όσων σήμερα πια έχουμε μάθει. Νομίζω κύριε Σαγητά κάπου θα πρέπει να γίνει μνήα, ίσως υπάρχει αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, να γίνει μνήα στην ε, επερχόμενη ε, αναθεώρηση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει πλήρως, να έχει μάλλον την πλήρη εξουσία να διεξαγάγει ε, έρευνες πλήρης και διαρκής ερευνητικές επιτροπές να μπορούν να συσταθούν στο Κοινοβούλιο. για την διαφάνεια και την σχέση αυτή με, την, ε, με το απόρριτο των εγγράφων. Για ένα υγιέ δημοκρατικό σύστημα πρέπει να υπάρχουν εδώ και κάποιοι έλεγχοι, κάποιε δοκιμέ. Είναι πολύ σχετικό ότι οι συνομιλίε για την αναθεώρηση της, του κανονισμού για τη διαφάνεια ακόμη δεν μπορούν να προχωρήσουν. Είναι μπλοκαρισμένε. Η επένδυση στην ασφάλεια στο διαδίκτυο στην επικοινωνία με τα τεχνολογικά μέσα. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να μας αποσχολήσει μετά τις εξελίξει των τελευταίων μηνών. Φάνηκε ότι είμαστε πολύ αφελείς και το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στην ασφάλεια των συστημάτων μας. Αλλά ευθύ εξ αρχή πρέπει να μα αποσχολήσουν τα συστήματα IT που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Έχουμε ήδη θέσει ερωτήσει και ακόμα. Με συγχωρείτε. Απαντήσεις περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Οι hacker ε, έχουν εχθρό την άλλη εβδομάδα, να το ξέρουν αν μας ακούνε. Δεν έχουμε... Εδώ μάλλον ήδη βλέπουμε ανακοινώσεις παντού στο κτίριο που λένε ότι δεν δουλεύει το wifi. Μα είναι γελίο, έτσι. Είναι γελίο. Αντί να βάζουμε χαρτιά που να λένε δεν έχει wi Wi-Fi, ίσως καλύτερα να στέλνουμε προσκλήσεις ε, στους ενδιαφερόμενους, όχι μόνο στους hacker, αλλά και στους εγκληματίες του διαδικτύου, να λέμε είναι ανοιχτές οι πόρτες μας, ελάτε. Μα σοβαρά τώρα, υπάρχουν εδώ ε, δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι που παίρνουν και πολλοί παχυλού μισθού, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συστήματο. Περιμένουμε τώρα απάντηση δύο μήνε μετά την παραβίαση. Εάν ήταν εδώ εταιρεία, αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν πεταχτεί στο δρόμο, θα ήταν απολυμμένοι. Γιατί το ανεχόμαστε αυτό, γιατί δεν έχουμε απάντηση για το σύστημά μα ακόμη δεν είναι ασφαλέ. Μπορεί να μου το, απαντήσει κανεί, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον εγώ θα φταίω. Και δύο τελικές παρατηρήσεις για, τον, για, την, για το δράση στους υπολογιστές σε νέφος, το υπολογιστικό νέφος, δεν συμφωνώ να προβλέψουμε ένα φραγμό, ένα φράχτη, τείχος προστασίας γύρω από το δικό μας σύστημα των υπολογιστών. Ένα ευρωπαϊκό διαδίκτυο, όχι, θέλουμε να είναι ανοιχτό αυτό για να μπορούν οι πολίτες να έχουν επιλογή και εταιρείε κίνητρο φτιάχνοντας καλύτερα συστήματα. Ασφαλέστερα. Καλύτερα συγκροτημένα. Δεν θυμάμαι τα λόγια ακριβώς ε, όπως τα είχε πει, αλλά ο κύριος εκείνος, ο γερμανός hacker που είχαμε εδώ και σε ακρόαση, έλεγε ότι εάν ε, κάτι πάει στραβά με ένα αυτοκίνητο που αγόρασε κανεί, είναι υπεύθυνο ο κατασκευαστή. Εμεί γιατί τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Και τελικά για το TGIT, ναι, Είμαι υπέρ της συμφωνία της Διατλαντικής για το ελεύθερο εμπόριο, αλλά τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να αποφασιστεί ή να προχωρήσει εάν δεν έχει αποσαφινιστεί η κατάσταση και δεν έχουμε σαφέστατες εγγύησεις για την προστασία των ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών μας από την άλλη πλευρά. Α, ανυπομονώ λοιπόν για τις μελλοντικέ συζητήσεις και ελπίζω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα ισχυρότατο πακέτο συστάσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, ο οποίος ε, μας ε, παρουσιάζει Μα υποβάλλει μάλλον μια πολύ καλή αφετηρία για τα συμπεράσματά μα. Πριν από έξι μήνε περίπου έκανε τι αποκαλύψει του Edward Snowden και είδαμε ότι όλο και περισσότερο το κράτος δικαίου, η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, των ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβαθμίζονται, χαλαρώνουν. Και πρέπει να πω ότι αυτή η χαλάρωση δεν γίνεται βέβαια γιατί υπάρχει ο Έντουαρτ Σνόντεν, ούτε και έκτοτε ξεκίνησε, απλά οφείλεται στις ε, δραστηριότητες και στα μέτρα και στην ομοθεσία που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις μας. Το αποκάλυψε με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος ε, ο Έντουαρτ Σνόντεν και νομίζω ότι αυτό πρέπει και εμείς στην έκθεσή μας να το αναφέρουμε ξεκάθαρα ζητώντας να αναγνωριστεί γι' αυτό που είναι ουσιαστικά ένας ε, άνθρωπος ο οποίος έδωσε πληροφορίες ουσιαστικά ε, για το πώς παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ιδιωτική σφαίρα των Ευρωπαίων πολιτών. Και καλό θα ήταν να το καλέσουμε και εδώ για να ακούσουμε τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει από πρώτο χέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα σχόλια της ηγετική των Ισκιωδών για την σημασία της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμφωνία πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για καλύτερη προστασία τη ιδιωτική σφαίρα ε, και των δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων πολιτών στη, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό συμπέρασμα αυτής της ε, ερευνητικής, της εξεταστικής διαδικασίας. Χρειάζεται και έλεγχος, χρειάζεται και εποπτεία. Όχι μια θολή έτσι, ε, μέτρα εποπτεία και από πλευράς είπα και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είδαμε με τις έρευνες που κάναμε ότι συνεχίζεται και εδώ στην Ευρώπη μια δραστηριότητα από τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών που έχει να κάνει με συνεργασία με τις αρχές των ΙΠΑ είτε με μαζικές παρακολουθήσεις ε, Ευρωπαίων πολιτών. Η εθνική ασφάλεια εξαιρείται, δεν υπάρχει κανένα έλεγχος, αλλά ακούσαμε και οι εκπροσώπου εθνικών κοινοβουλίων. Ούτε και σε εθνικό επίπεδο κατάλαβα να υπάρχει επαρκή έλεγχο. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε και θα πρέπει να υπάρχουν ε, κανόνε ε, για τη δράση των ε, υπηρεσιών πληροφοριών των χώρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πρέπει να πούμε ότι και επιβολή δεν υπάρχει, είναι φυσικό αυτό, από τι αστυνομικέ αρχέ ή άλλε αρχέ που είναι αρμόδιε για το θέμα αυτό, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν έχουμε κυβερνοεπιθέσει από αρχές τρίτων χωρών ή από εταιρείε τρίτων χωρών ή και από εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ευρώπη και αυτέ οι επιθέσει γίνονται ε, στου διακομιστέ και τα συστήματα φορέων παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Βλέπουμε ότι επανειλημμένω ε, η Ευρώπη ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει έτοιμο από καμία εθνική αρχή ακόμη και για να ερευνηθούν οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές. Είναι γελίο και σκανδαλώδες κάτι τέτοιο. Να έχουμε τέτοια έλλειψη επιβολής του νόμου, τεράστια έλλειψη επιβολής του νόμου. Πρόσφατα μόλις εγκρίναμε, μόνο εγκρίναμε κανόνες για την επιβολή ε, του νόμου σε ό,τι αφορά τον κυβερνοχώρο, πρέπει να εμείνουμε στην εφαρμογή αυτών των κανόνων. Επίσης θέλω να πω ότι και το θέμα της ευθύνης είναι σημαντικό για τα συστήματα που παρέχουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες στην ψηφιοποιημένη κοινωνία που ζούμε. Αντί να επιδοτήσουμε την ε, παραβίαση κρυπτογράφησης και την παραβίαση αυτών των συστημάτων θα πρέπει να επενδύσουμε στην ανωνυμοποίηση και στην κρυπτογράφηση, ώστε να μπορεί ο πολίτης ε, να προστατευθεί και να διαφυλάξει την ιδιωτική του σφαίρα εφόσον το επιθυμεί. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα και αυτό πρέπει να ενισχυθεί και εδώ στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια θα πρέπει να δώσουμε και ένα θετικό παράδειγμα σε Ευρώπη. Ε, ε, reference to the... Και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι στην έκθεση υπάρχει αναφορά ε, την ε, παρακράτηση γενικώ όλων των στοιχείων κάποιου ατόμου που μπορεί να μην είναι υποπτό. Blanket retention. Αυτή η οδηγία ε, της Ένωσης για την παρακράτηση στοιχείων αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Η Φύλαξη των στοιχείων, παραδείγματο χάρη των στοιχείων επιβατών, το PNR. Πολλοί λένε θα σώσει, ε, θα αυξήσει την ασφάλειά μα, θα προστατεύσει. Όχι, αυτό είναι λάθο. Παραβιάζονται με τον τρόπο αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να χαράξουμε μια γραμμή μεταξύ του τι είναι αποδεκτό σε επίπεδο ελέγχου, εποπτείας, στις κοινωνίες ό,τι αφορά τα στοιχεία και την επικοινωνία και μεταξύ του τι δεν είναι αποδεκτό. Επίσης θα πρέπει να επεξεργαστούμε αποτελεσματικού μηχανισμούς εποπτείας και αυτό πρέπει να το κάνουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξαρτήτως ε, του τι λένε οι εθνικές μας κυβερνήσεις, διότι σε, εθνική, σε έξι μήνες δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με το σωστό τρόπο τις αποκαλύψεις. Ε, είδαμε μάλλον σε αυτούς τους έξι μήνες δεν ήταν ικανεί να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αποκαλύψεις και έχουμε και εκλογές το Μάιο. Θέλουμε να δω, εμείς να δώσουμε το στίγμα μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ λοιπόν πρόεδρος, κύριε Έρνστ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο είναι φιλοφρόνηση. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο γιατί μπόρεσε να φέρει σε πέρα σε ένα τόσο δύσκολο έργο και έχει συνεργαστεί με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους εμπλεκομένους. Αν δούμε λοιπόν το, την έκθεση αυτή ως σύνορο, είναι φανερό ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το πιο δύσκολο ίσω όλης αυτής της θητείας για πάρα πολλούς ε, λόγους. Πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει μια πλήρης εικόνα της γενικότερης προβληματικής. Προφανώς αναφέρεται η απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και Αμερικανινών αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θεσμικά και νομικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένη αυτή η προβληματική όπως θέλησαμε να το τονίσουμε γιατί πρόκειται για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερία, ελευθερία του έκφρασης, ελευθερία επικοινωνίας, ελευθερία του τύπου και όλα αυτά. Και εμείς φυσικά έχουμε περιοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνά μας υπάρχει και το επίπεδο του τι γίνεται μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν είμαστε απόλυτα αθώοι για τα θέματα αυτά, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντίστοιχε ενέργειες παρακολούθησης και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι προσκάλεσε παραγωγικά τη Γερμανίδα Καγκελάριο ο Ομπάμα αλλά δεν βλέπουμε όλα αυτά να οδηγούν σε κάποια κίνηση στις χώρες μας και θα έπρεπε να υπάρχουν ενέργειες και προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω δυσκολίες σε σχέση με θέματα νομικού χαρακτήρα. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς ενός που δεν είναι Αμερικάνος στις ΗΠΑ και πώς μπορεί να διεκδικήσει τα νομικά του δικαιώματα είναι απόντα αυτά τα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με το επιχείρημα της προστασίας της εθνικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι πού φτάνει η ασφάλεια, η εθνική, η ευρωπαϊκή, όλα αυτά, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και ξέρουμε ότι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κανείς να τα δικαιολογήσει όλα με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην έρευνα αυτή που δεν νομίζω ότι το, το διεξήλθαμε τελείω. Και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο στο να καταργηθούν οι διατάξεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και εδώ θα πρέπει να δούμε αν πράγματι είναι τόσο σημαντική η ασφάλεια ώστε να πρέπει να υπερκεράσει όλες τις ε, ελευθερίες. Εμείς ως ομάδα της αριστεράς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η έκταση έχει πολλά πράγματα τα οποία τα τονίσαμε εμείς και τα οποία προήλθανε και από τις ακροάσεις που κάναμε. Ανεξάρτητα από όλα αυτά όμως, είναι πολλά στοιχεία τα οποία έχουν μείνει απ' έξω. Πολλές συστάσεις και πολλές ε, διαπιστώσεις για μένα είναι απόλυτα απαραίτητο να μην συνεχιστεί η εφαρμογή του Safe Harbor στην τωρινή μορφή του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να στα, να, να, δεν μπορούν να σταθούν τα επιχειρηματά μας όταν αποδεχόμαστε να υπάρχει παραβίαση των συνθήκων που έχουμε συνάψει ήδη. Και αυτή τη στιγμή παραβιάζονται αυτά τα συμβατικά στοιχεία της, των συνθήκων. Το ίδιο πράγμα ισχύει με το ΣΟΥΙΦ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία στην τωρική της μορφή. Δεν είναι επαρκής οι ρυθμίσεις με την ε, κατάσταση του SWIFT. Και είναι τώρα κάτι το οποίο μου φαίνεται πεδαριώδες να συνάπτουμε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και να διαπραγματευόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. Νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση και χωρίς πίεση δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά για να εξασφαλίσουμε ότι Εάν υπάρξει μια συμφωνία θα πρέπει να είναι μια ικανοποιητική συμφωνία. Θα πρέπει ακόμα και αυτή τη συμφωνία λοιπόν του διατλαντικού εμπορίου να την παγώσουμε μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες να εξασφαλίσουν μια σωστή διαδικασία προστασίας δεδομένων. Επίσης η προστασία των καταγγελόντων είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό είναι ένα στοιχείο τη έκθεση, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να υλοποιηθεί σε, νομικό, σε νομοθετικό επίπεδο φυσικά πρέπει να ενσωματωθεί και στην νομοθεσία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ελέγχεται επίσης ότι υπάρχει τεχνολογική αδυναμία της Ευρώπης για τα θέματα αυτά της πληροφορικής. Μα το θέμα είναι που βάζουμε εμείς την προτεραιότητά μας. Για μένα η προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία των δεδομένων και των ελευθεριών των προϊόν, των πολιτών. Εγώ θέλω τώρα να πω κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να θέσουμε και το ερώτημα τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούν οι μυστικές υπηρεσίες. Είναι αναλογική η δράση τους σε σχέση με τους στόχους που εξυπηρετούν. Ποιος είναι ο στόχος αυτών των μυστικών διπλωματικών ενεργειών. Κανεί δεν θέτει αυτό το ερώτημα. Εγώ δεν νομίζω ότι αρκεί το να παραγνωρίζουμε αυτό το θέμα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις μυστικές συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα ανεξάρτητο φορέα ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι μονάχα οι φιλικές συνομιλίες που κάνουμε με προσώπους των μυστικών υπηρεσιών σε μια επιτροπή πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες να εφαρμόσουμε έλεγχο. Και αυτό πρέπει να ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά παραθυράκια, πολλές τρύπες αναφέρθηκα ήδη στις αντιτρομοκρατικέ νομοθεσίε, και επιπλέον πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να δαπανίσει και περισσότερα ποσά και να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την δική του ασφάλεια σε επίπεδο κυβερνοχώρου. Και το ερώτημα είναι αν φτάνουν όλα αυτά. Μπορούμε πράγματι να πάμε στην πηγή του προβλήματος. Κάνουμε κάτι το οποίο θα θέσει την μαζική παρακολούθηση πράγματι ένα αμφιβόλο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ε, απαντήσω. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ωραία, κάναμε αυτή την έκθεση, τη δημοσιεύουμε, θα την κοιτάξει η Κομισιόν και τι θα προέλθει από όλα αυτά. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. πρέπει να αρθρώσουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες μας σε αυτό το τομέα, ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει και αυτό σημαίνει και συμφωνία των κρατών μελών. Νομίζω ήμουν ιδιαίτερα γενναιόδορη με τους κέντρους εισηγητές και θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρή με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να με συγχωρείτε. Το λόγο έχουν τώρα οι συνάδελφοι που θέλουν να, ε, να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Πίπερ, η κυρία Λάτφορτ, η κυρία Γκόμες, η κυρία Σαρχιντίνη, η κυρία και ο κύριος Έντσου. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να προσθεθεί, το λόγο έχει ο κύριος... Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πύρκα. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις και μετά θα προχωρήσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία για, για ε, συγκεκριμένα ερωτήματα. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μωράες για την πληρότητα και την ε, ε εξονυχιστική μορφή της έκθεσής του υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία προέρχονται από εμπειρογνώμονες και τα οποία θα πρέπει να είναι και η βάση της περαιτέρω ε, βάση των ενεργειών μας και γνωρίζουμε ότι και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ υπάρχει μια σειρά ενεργειών από Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές που θεωρούν ότι δεν εφαρμόζεται πάντα η νομοθεσία των ΗΠΑ, ούτε και εκεί. Υπάρχουν απόλυτα δικαιολογημένες κριτικές που αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Αλλά υπάρχουν και κάποιες υπερβολικές διατυπώσεις και κάποιοι, ε, κάποιες ε, επιθυμίες που διατυπώνονται όπως αυτές στο άρθρο 21 που ζητούν από τα κράτη-μέλη να μην επιτρέψουν δραστηριότητες κατασκοπίας άλλων χωρών στις χώρες τους. Όλα αυτά βέβαια φαίνονται κάπως αφελή, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά να μπορέσει κανείς να τα υλοποιήσει. Ίσως εδώ λοιπόν θα πρέπει να μην περιλαμβάνονται τέτοιες διατυπώσεις στην έκθεση. Υπάρχουν και άλλες αιτήσει οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εξασφαλίζουμε ότι τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Τι γίνεται όταν υπάρχει κάποια α, κάποια αγωγή εναντίον των συμφωνιών αυτών, ε, τι γίνεται και πώς εξασφαλίσουμε την διατήρηση του ρόλου τους. Έχουμε λοιπόν πολλές σημαντικές ε, ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να επαναφερθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών για να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και η εμπορική συνεργασία ΗΠΑ και επίσης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα βρούμε τα απαραίτητα μέσα για να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, είτε είναι τα συμφέροντα των πολιτών, είτε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Εδώ μια πρώτη διεκδίκηση που όλοι υπεστηρίζουμε όλοι είναι να ότι θα πρέπει να έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα για τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης όπως αυτών των Αμερικανών Δεύτερον, να υπάρξει μια συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Και ένα τρίτο που είναι πολύ σημαντικό για μένα, θα πρέπει με σαφέστερο τρόπο από ό,τι στην ε, έκθεση αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δική της υπηρεσία αντικατασκοπίας. Χρειαζόμαστε όχι μια υπηρεσία ευρωπαϊκής κατασκοπίας αλλά αντικατασκοπίας για να μπορέσει να προστατεύσει τα εμπορικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιριών από ξένες παρεμβάσεις και προσπάθειες κατασκοπίας. Όλα φυσικά αυτά πρέπει να γίνονται κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου κοινοβουλευτικού και επί τη βάση συγκεκριμένων κανόνων. Θα ήθελα λοιπόν να αναλυθούν όλα αυτά τα στοιχεία για που θα οδηγήσουν σε καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών μέσα σε μια πολύμερη συμφωνία. Αυτό δεν απαιτεί καμία αλλαγή των συνδικών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε πολυμερές επίπεδο, να καθοριστούν οι κανόνες οι οποίοι, οι οποίοι διέπουν την ε, ασφάλεια των ε, ανταλλαγών πληροφοριών και εξασφαλίζουν και τον έλεγχο τους. Στα σημεία 65 και 66 ο κύριος Μωράης έχει αναφερθεί στο σημείο αυτό, αλλά θα ήθελα να υπάρξει και περαιτέρω διευκρίνηση και αποσαφήνιση για τα θέματα αυτά για να υπάρξει και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών και φυσικά πρέπει να βελτιωθεί και η ανεξαρτησία σε επίπεδο πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ εμείς έχουμε το υπολογιστικό δίκτυο, πρέπει να έχουμε ένα υπολογιστικό δίκτυο που να είναι ελέγξιμο από εμά, πρέπει οι διακομιστές να είναι ελέγξιμοι για να μπορούμε να ελέγχουμε πού πηγαίνουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ κύριε Λάτφορτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φοβούμαι ότι θα κάνω τα σχόλιά μου βιαστικά με κάποια γένεια και θα αναγκαστώ να φύγω τρέχοντας μετά γιατί πρέπει να λείψω. Ε, η Σόφη μας είπε ότι πρέπει να βάλουμε ένα, φράχτη γύρω από το ευρωπαϊκό διαδίκτυο, ένα φραγμό. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ακριβώς, διότι ανεξαρτησία θα πρέπει να υπάρχει στο ευρωπαϊκό διαδίκτυο και στα, στις υπηρεσίες νέφους ε, θα πρέπει να προσέξουμε ε, μήπως χρειάζεται ένα τέτοιο τείχος προστασίας. Τώρα γιατί, ε, για την ανεξαρτησία θα πρέπει να προσέξουμε πώ θα χρησιμοποιούμε τον όρο, πώ τον χρησιμοποιήσει και πρόεδρο Ρέντινγκ. Και νομίζω ότι καλά θα ήταν και αυτέ τι αναφορέ να έχουμε υπόψη μα, θα μα χρησιμεύαν. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε αντιφάσει στην έκθεση, διότι συμφωνώ κατά μεγάλο μέρο ότι η συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσε να εξαρτηθεί από πολλά στοιχεία, αλλά ένα από αυτά, το βασικότερο ίσως, θα ήταν η εμπιστοσύνη στο επιγραμμικό περιβάλλον. Να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τις ΗΠΑ που, έχει, που έχουν προβλήματα οι αναταράξεις, αλλά και η Ευρώπη. Και το βρίσκω κάπως ε, περίεργο να ζητούμε τώρα την άρση του ασφαλούς λιμένος. Όταν ε, στη λογική σκέψη λέγεται ότι ή φαίνεται να υπάρχει μια ευνοϊκή μνήμα για το γεγονό ότι η Επιτροπή έχει απευθύνει κάποιε συστάσεις προ τι ΗΠΑ και πρόκειται μέχρι το καλοκαίρι του 2014 να εξεύρουν από κοινού τα ενδικά μέσα που θα πρέπει να ασκηθούν σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υπάρξει ανάκληση τη ρήτρας για τον ασφαλή λιμένα. Και η FDC έχει παραδεχτεί ότι ο ασφαλής λιμένας θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ώστε να βελτιωθεί η διάσταση του μέτρου. Το θέμα λοιπόν είναι εάν μπορεί κανείς να έχει πραγματικές εγγύσει ή δικλείδες ασφαλεία, και το βρίσκω λίγο περίεργο να σημειώνουμε ότι η διαδικασία υπάρχει για τον ασφαλή λιμένα αλλά να ζητάμε από μόνοι μα την άρση αυτομάτω τώρα δέχομαι ότι είστε πρόεδρο τη ε, αντιπροσωπεία για τι σχέσει με τι ΗΠΑ. Θα με ενδιαφέρε ιδιαίτερο να υπάρχει ένα ενίο οικονομικό χώρο, όχι αφελώ, χωρί να ξεχνάω όλε τι υπόλοιπε προκλήσει που τίθενται, ε, ούτε για το επιγραμμικό περιβάλλον, αλλά πραγματικά κάπω ε, δεν αισθάνομαι άνετα με την τόσο προφανή αντίφαση που υπάρχει εδώ. Δηλαδή, άρση τώρα, αλλά με ανοιχτή διαδικασία αναθεώρηση και ενδεχομένω βελτίωση τη ρήτρα για τα ασφαλή Δεν μου αυτό. Ευχαριστούμε, λέτε Λάτφορντ. Κύριε Μωράη, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι πριν φύγει η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ, Κίνκα. Με συγχωρείτε που καθυστερώ. Απλώ πριν φύγει η κυρία Λάτφορντ και για την ε, σοφή και το cloud computing. Στι παρατηρήσει μου και στο κείμενο τη έκθεση, νομίζω ότι δεν είναι πολύ σαφέ το πώ εκφράστηκα για το cloud computing. Ίσως να το αποσυμφωνήσουμε. Ναι, θα χρειαστεί ένα τείχος προστασίας, ε, αλλά και η πράσπιση της ανεξαρτησίας μας. Δεν είμαι θειασότης της ε, απομόνωσης του ε, ευρωπαϊκού νέφους, των υπηρεσιών νέφους, γιατί μας κοιτάζουν και οι πολίτες και το κοινό, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Το λέω λοιπόν τώρα γιατί δεν θέλω να μείνει να πάρει το... και να έχει φύγει η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μωράης. Η κυρία Γκόμες. Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Κλοντ Μωράης για την εντατική και υψηλής πρόταση έκθεση που μας έχει υποβάλει. Μετά από όλες τις ακροάσεις, συνομιλίες και επαφές που είχαμε. Εξαιρετική βάση για τη δουλειά μας, αλλά ακόμη περισσότερο ως συνεισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την ε, νομοθέτηση αυτή, πραγματικά χαίρομαι για τον τρόπο που ενσωματώθηκαν οι απόψεις μας, ε, όπως τόνισαν και ο κύριος Αλαφράκα και ο κύριος Μωράης. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τις κοινέ αξίες, τις κοινέ μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες αξίες. Νομίζω ότι αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό για ανθρώπους που έρχονται από πρώην ολοκληρωτικά καθεστώτα. Εγώ έζησα 21 χρόνια κατά από δεκατορικό καθεστώς. Οπότε δεν είναι θέμα το μόνο θέμα το κράτος δικαίου απλώς ή ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου των πολιτών απλώς, αλλά το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Και εδώ πραγματικά πιστεύω ακράτατα, ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν ανατρέχουμε διαρκώ την ίδια μοθολογία που χρησιμοποιούν και οι τρομοκράτες. Έτσι είναι η δημοκρατική και νόμιμη μεθοδολογία. Δεν είναι αποτελεσματικό τρόπο καταπολεμήση τη τρομοκρατίας αυτός. Όχι. Πρέπει να ενισχύσουμε πρέπει να καταπολεμήσουμε του τρομοκράτε, αλλά όχι με το να γίνουμε εμεί οι ίδιοι τρομοκράτε. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι το σημαντικό είναι όχι απλώς να δίνουμε πληροφορίες για τον τρόπο που ο ιδιωτικό βίο των πολιτών της Ευρωπαϊκή Ένωση ή των ΗΠΑ παραβιάζονται κατάφορα, αλλά και για το πώς αυτό έχει παρακαμφθεί για σκοπούς όχι και τόσο πολύ οργουελικούς για την πολιτική κατασκοπία και ούτω καθεξής, αλλά ακόμα χειρότερα για τον τρόπο που έχει φανεί ότι εργαλεία τα οποία αρχικά έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν είναι αποτελεσματικά. Διότι αν το σύστημα μαζικής παρακολούθησης που χρησιμοποιήσει η NSA υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της δημοκρατίας έχει διαστρεβλωθεί και έχουν καταβληθεί για αυτό τόσα κονδύλια, έχουν ε, αναλωθεί τόσοι πόροι για την μαζική των πολιτών όλου του κόσμου και έχει επιτραπεί σε δύο Τσετσένους να βάλουν βόμβες στον μαραθώνιο της ε, Βοστόνης ε, είναι σαφές ότι η διάσταση των μυστικών πληροφοριών δεν λειτουργήσε. Υπάρχει αναποτελεσματικότητα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν όντως ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και κατά πολλούς τρόπους καλύπτεται. Πιστεύω ότι έχουμε μεν ισχυρή προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν εφαρμόζεται. Έχουμε πρόβλημα επιβολή, όπω είπε η Σοφή. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταγορούμε τι ΗΠΑ. Οι δικέ μα υπηρεσίε φταίνε, οι δικοί μα φορεί, τα δικά μα θεσμικά όργανα που δεν εκτελούν το ρόλο τη εποπτεία που ε, του έχει ανατεθεί. Πολιτικό, ε, πολιτική, ε, δικαστική, οποιασδήποτε εποπτεία, όπω με την Belgacom. Δεν είναι ευθύνη των ΗΠΑ αυτή, ένα ευρωπαϊκό κράτος ευθύνεται. Και δεν είναι μόνο η Belgacom. Δεν είναι μόνο άσχετοι ευρωβουλευτές που μπορεί να φταίνε. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο κύριος Μπαρόζο, ο κύριος ε, Μπαρνιέ, ο κύριος Ρέντινγκ που μπορεί να είναι θύματα κατασκοπίας. Σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ έχει διοργανωθεί συζήτηση για το αν η NSA κατασκόπευσε μέλη του Κογκρέσου και δεν το αρνήθηκε ακόμα η NSA. Τι άλλο πια θα γίνει. Όταν είχαμε τορμοκατηθεί με τις αποκαλύψεις που περιμέναμε ακόμα από τον Σνόντεν, λέγαμε τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Γιατί τότε ήδη ξέραμε για την κατασκοπία της Μέρκελ. Ε, μπορεί να έχουν κατασκοπεύσει και τον Ομπάμα τον ίδιο. Ε, και το, το απίστευτο είναι ότι κανείς δεν το έχει αρνηθεί ακόμα. Κανείς δεν βγήκε να πει «ε τίποτα». Οπότε εδώ μιλάμε για την ουσία του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, του δημοκρατικού καθεστώτος. Ε, κλείνοντας, να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες των υπολείπων ε, για την ε, διατύπωση του άρθρου 59. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάπως η διατύπωση της πρότασης αυτής, διότι ακριβώς για την ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνη όπως το θέσατε. Το πιο ενδιαφέρον είναι κατά την άποψή μου οι Ηνωμένε Πολιτείε να συμμετέχουν στον οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι που μπορεί να πλήξει τη συμφωνία ομπρέλα, την ε, σφαιρική αυτή συμφωνία. Πώ θα οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνη, εάν βασικά δικαιώματα άσκηση, προσφυγή σε διοικητικό και, δικαστικό επίπεδο ε, δεν επιτραπεί σε Ευρωπαίου πολίτε για τι ΗΠΑ. Και ακόμη οι ευθύνε εποπτεία. Αυτό είναι ζωτικό ρόλο που δεν μπορούν να έχουν μόνο τα εθνικά κοινοβούλια. Άμα δεν κάνουν τη δουλειά του, οφείλουμε και θα πρέπει να αντιστρέψουμε τη αρχή τη επικουρικότητα. Μια αντίστροφη επικουρικότητα. Άμα δεν κάνουν τη δουλειά του, όπω πολλοί κάνουν, δεν κάνουν μάλλον, δηλαδή στη χώρα μου πρώτη-πρώτη, την Πορτογαλία, ε, τότε αυτό το κοινοβούλιο, το δικό μας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες των κρατών μελών εκτελούνται σωστά. Ευχαριστούμε, κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, και Χιμένεθ Μπεθερή. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Μωράης. Είχαμε συνεργαστεί και στην επίσκεψή μας ε, στη Ουάσιγκτον όπου και παληθεύσαμε επί τόπου ότι αυτό το θέμα δεν ανησυχεί και ενδιαφέρει μόνο από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και την αμερικανική σε σχέση με την Ευρώπη και αυτό είναι κάτι θετικό γιατί δεν ήθιστε να ενδιαφέρονται οι Αμερικάνοι πάρα πολύ για ε, διάφορα θέματα που μας αφορούν. Αυτή τη φορά όμως ε, συνέβη αυτό. Υπάρχουν ζητήματα που μας ε, ενδιαφέρουν και μας ανησυχούν εδώ στο Κοινοβούλιο καθότι είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών οι πολίτες ενδιαφέρονται για την ιδιωτική σφαίρα αλλά και για την ασφάλειά τους. Ε, και εμείς το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θα ε, ασχοληθούμε με ό,τι έχει να κάνει με την τρομοκρατία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ε, απαράδεκτες οι μαζικές αυτές παρακολουθήσεις είναι καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά η αναστολή των προγραμμάτων συνεργασίας για την καταπολέμηση της αποκρατίας ε, δεν είναι λύση. Το SWIFT για ποιο λόγο πρέπει να γίνει ο Πομπέος τράγος αυτού του σκανδάλου που επαναλαμβάνω ότι είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να τον εχθούμε. Το SWIFT δεν έχει άμεση σχέση με την κατασκοπία, με τις μαζικές αυτές παρακολουθήσεις και είναι τη πάση γνωστό ότι μέχρι στιγμή λειτουργούσε πολύ καλά. Η επίσκεψή μα λοιπόν ε, στις ΗΠΑ, στη Ουάσιγκτον και μπορεί να το ε, επιβεβαιώσει και ο Κλοντ Μωράης, ε, απέδειξε ότι σε περιπτώσει ψηλού κινδύνου είμαστε αποτελεσματικοί. Βέβαια δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για προφανείς λόγους ε, οι διάφορες τρομοκρατικές Ενέργειε που απεφέχθησαν λόγω αυτή τη πολύ αποτελεσματική εργασία, ήταν όμω εκατοντάδε. Θα πρέπει να σα πω, συμφωνώ και με τον Άξελ Βό, τον σκιώδη συγκητή για το ότι θα πρέπει ε, την ΕΝΙΣΑ, το EU, τη Europol, ε, όλες τους ευρωπαϊκούς αυτούς οργανισμούς να τους ενισχύσουμε και να έχουμε και ίσως και έναν οργανισμό αρμόδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είμαστε πιο αυτόνομοι και να έχουμε και καλύτερη συνεργασία με τις ΕΠΑ. Πάντως σημαντικό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους ε, πολίτες να είμαστε ένα ισχυρό κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να δείξουμε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα, τα είπε και η κυρία Ιντβέλτ. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ευθύνης, πευθυνότητας και δεν θα ήταν υπεύθυνο να αναστείλουμε το ε, SWIFT, διότι μόνο όσοι χρηματοδοτούν ε, την τρομοκρατία ε, θα χαρούν με κάτι τέτοιο. Στηρίζω το κείμενο, αλλά όπως είπα έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντσου. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Κλοντ Μωράης για την έκθεσή του. Αλλά να τον συγχαρώ και για το πνεύμα συνεργασίας. Και γιατί υπήρξε άκρος εργατικός, με εντυπωσίαση η εργατικότητά του. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα της έκθεσης, πάντως θεωρώ ότι όταν εγκριθεί αυτή η έκθεση και με τις ε, πετούμενες τροπολογίες βέβαια, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινητοποιηθεί θα πρέπει να κινητοποιηθεί ώστε αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος, η δημοκρατική αυτή εποπτεία να επιβληθεί για να αποτραπούν μαζικές παρακολουθήσεις στο μέλλον. Πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ καταπολέμησης τρομοκρατίας αφενός και καταχρήσεων που είδαμε μέχρι τώρα αφετέρου. Θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι που έγινε στη Ρουμανία, τη χώρα πριν από κάποιες ημέρες. Ο κεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών ε, στη Ρουμανία έπεσε θύμα ε, πειρατείας, hacking, ναι. τα προσωπικά του, και προσωπικοί του λογαριασμοί παραβιάστηκαν. Άρα θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω πράγματα για να ενισχύσουμε την προστασία. Αυτά είναι η ανεκδότη λοιπόν. Πρόεδρο, ναι παρακαλώ, επόμενα είστε πολύ σύντομοι. Α, ο κύριος Μωράη. Σύντομο θα είμαι, Κίνγκαλ. Πόσο σύντομο θε να είμαι. Πάρα πολύ σύντομο. Για να είμαι ειλικρινή, Αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι υπάρχει μεταξύ των μελών τη Επιτροπή μα, υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνη και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εμπειρογνώμονε στα θέματα ε, ε προστασία δεδομένων και εγώ δεν ήμουν εμπειρογνώμων στα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι φανερό από τις παρεμβάσεις τους υπάρχουν ε, άτομα που είναι ειδικοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε άλλους τομείς και το είδατε αυτό από τις ε, συνεισφορές τους δεν θα απαντήσω λοιπόν ερωτήματα όταν ήταν ουσιαστικά σχόλια απλώς να σταθώ σε ορισμένα σημεία όπου οι συνάδελφοι μου ζήτησαν να δώσω μια απάντηση. Και για την Τερέζα και για τον κύριο Πέρκερ, για να μην μου πει κανείς ότι δεν απάντησε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα, δείξατε το ζήτημα της συλλογή πληροφοριών και του SWIFT. Θέλω να πω τελείως σαφώς ότι θα υπάρξουν στοιχεία και στην τελική έκθεση. Εδώ είναι απλώς το σχέδιο έκθεσης και είχαμε μια πολύ έντονη δραστηριότητα για τα θέματα όπως το SWIFT, το Safe Harbor, στο παρελθόν, με ψηφίσματα, με δηλώσεις της Επιτροπής κτλ. Υπήρξαν πολιτικές δυσκολίες και διαφορές μεταξύ των ομάδων μας και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να ανταρακλώνται στην τελική έκθεση. Θέλω να κατανοήσουν οι συνάδελφοι ότι κατανοώ γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζω τη σημασία που έχει η συμφωνία SWIFT. Ήμουν παρόν όταν έγινε η διαπραγματεύση αυτή τη συμφωνία. Αυτό το πρέπει να κάνουμε όμω στην έκθεση είναι να δούμε τις ίδιες αυτές τι καταγγελίες αλλά μπορεί να προκύψουν διαφορετικέ απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε σχέση με το περιεχόμενο της έκθεσης. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι κάποιε από αυτές τι δυσκολίε και διαφορε θα αναφέρονται. Επίση, οι παράγραφοι τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που αναφέρθηκαν από τον κύριο Σαλαφράγκα ενδεχόμενε ε, τροπολογίες και αυτό αναφέρθηκε και από την κυρία Γκόμες. Ελπίζω ότι αυτές οι τροπολογίες δεν θα αλλάξουν την βασική γραμμή και έμφαση της έκθεσης που αντανακλούν τη θέση των σκιώδων εισηγητών. Είναι κοινοτυπία το να ευχαριστήκαν οι του Αλλά θέλω να πω ότι εδώ οι σκιοδησηγητέ δημιούργησαν αυτή την έκθεση μέσω των εγγράφων εργασίες του. Αυτή ήταν η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Αυτό που θα ελπίσω είναι ότι αν δει σε αυτή την έκθεση, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλη τη γραμματεία για το έργο το οποίο έφερε σε πέρας. Αν δείτε τις σελίδες 32 και 33, Υπάρχει αυτή η έννοια του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Χαμπέας Κόρπους που είναι μια απάντηση ουσιαστικά στην κυρία Ένς, δεν ξέρω αν η Κορνηλία είναι ακόμα στην αίθουσα. Εντάξει, να επιταχύνω. Ρώτησε τι θα γίνει σε την έκθεση, αν θα την πετάξουμε μετά στα σκουπίδια, μετά τους επένους. Και υπάρχει πραγματικά ένα χρονοδιάγραμμα για τις συστάσεις αυτές και τη συνέχιση αυτή τη έκθεση Λόγω πίεση χρόνου θέλω να σταθώ μονάχα σε αυτό το σημείο. Αυτό το οποίο γίνεται στην έκθεση αυτή και πώ θα ε, αναπτυχθούν περισσότερα αυτά τα ζητήματα έχει να κάνει με δύο σειρέ θεμάτων. Και επειδή δεν είμαι εμπειρογνώμων όπω είναι πολλοί συνάδελφοι, υπάρχουν από τη μία πλευρά οι τομεί όπου έχουμε πραγματική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και άλλες που δεν έχουμε, αλλά έχουμε μια ηθική ευθύνη. Έχουμε λοιπόν εκεί πολιτική και ηθική ευθύνη, διότι προερχόμαστε από τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και μας ρωτάνε οι πολίτες μας τι κάνουμε για τα θέματα αυτά. Αλλά εκεί που έχουμε αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διαπραγμάτευσης για το Safe Harbor, για το SWIFT κτλ. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα και ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης εστιάζει σε αυτό το ψηφιακό habeas corpus, ώστε και η Κομισιόν αλλά και τα κρατη να μπορούν να δώσουν συνέχεια. Δεν μπορούμε εμείς να παραγνωρίσουμε την ε, ανάγκη να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη στους μηχανισμούς εποπτείας δεν θέλουμε να αποσύσουμε τις δικές μας ευθύνες, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι υπάρχουν θέματα στην αρμοδιότητα των κρατών μερών. Όταν φτάσουμε σε αυτά τα θέματα που είναι σαφής η αρμοδιότητα, όπως είναι το SWIFT, Safe Harbor κτλ, ακόμα και εκεί που υπάρχει διαφορά απόψεων, θα πρέπει να μπούμε σε αυτό το χώρο και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σαφή σύσταση όταν φτάσουμε στο επίπεδο των τροπολογιών και όταν ψηφιστούν και καταλήξουμε σε μια ενιαία άποψη. Με την έκθεση αυτή λοιπόν που να γίνει σαφές ότι είμαστε ένα σοβαρό κοινοβούλιο. Διάβασα αυτή την βδομάδα στον Economist μια στήλη του ανταποκριτή του Economist στην Washington που ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εξοργισμένο και παραδέχτηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Είπε ότι είναι πολύ καλή στο να εξοργίζονται αλλά όχι τίποτα άλλο. Όπως είπε και η Σόφι Ίντφελτ, θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί υπάρχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιμετώπισαν όλες αυτές τις 15 ακροάσεις που ήταν πολυτεχνικές. Υπήρξαν τα μέλη αυτά που πήγαν στη Ουάσιγκτον, υπήρχαν ισχυώδεις συγητές που βοήθησαν. Δεν είδα ποτέ σε μια έκθεση να υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη, διάχυτη και νεφελώδη διαδικασία και να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη και λεπτομεριακή έκθεση. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι συμμεριζόσαστε την χαρά μου που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάτι που δεν είναι απλώς οργή, αλλά μία σειρά από συγκεκριμένες συστάσεις και ελπίζω θα το δείτε αυτό όταν φτάσουμε στο στάδιο των ε, τροπολογιών και θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και περιμένω για τις επόμενες εβδομάδες τις δικές σας ε, συνεισφορές και ευχαριστώ την Γίγκα για την συνεργασία της. Πρόθεσμη για τις τροπολογίες είναι 22 Ιανουαρίου, 6 η ώρα το απόγευμα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι για τη συνεργασία σας. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο στη μέση διαταξή μας για αυτό το απόγευμα. η παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης του κ. Σαλαμπάν προς την Επιτροπή Ήτρε, όπου είναι αρμόδια η κυρία Πιλά Δεκαστήγιο, πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και δίνω το λόγο αμέσως στον εισηγητή ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ιδίως μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημαντική συζήτηση ε, του εγγράφου του κυρίου Μωράης Είχα την ε, δυνατότητα να είμαι και εγώ στην Ουάσιγκτον ε, ως μέρος της αντιπροσωπείας και με βοήθησε στο να συντάξω και το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Για την εσωτερική αγορά ηλεκτρονικών κοινωνιών. Θέλουμε να έχουμε μια ενιαία ανταγωνιστική αγορά στον τομέα των ηλεκτρονικών κοινωνιών. Αυτό είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πλευρά καταναλωτών σε ό,τι αφορά το σεβασμό στα δόντια προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών της πληροφοριών. Χαιρετίζω λοιπόν την προσπάθεια της Κομισιόν να διευκολύνει την εναρμόνιση των ε, δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. Έχουμε λοιπόν την ηχεμήθεια ε, της επικοινωνίας, η ιδιωτική σφαίρα, τα προσωπικά δεδομένα είναι επίσης πολύ σημαντικά για να ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη η καταναλωτέ. Και μόνο έτσι θα πετύχει αυτή η στρατηγική. Θα πρέπει οι καταναλωτέ να είναι βέβαιοι ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους όποτε χρησιμοποιούν τις υπηρεσίε και τα δίκτυα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Και κάθε ε, παραβίαση των δικαιωμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτή η γνωμοδότηση εστιάζει στις πτυχές της πρότασης που θα επηρεάσουν κατά πάσα πιθανότητα προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη, τα περιοδική σφαίρα ή την εχεμήθεια, το απόρριτο των επικοινωνιών, κεφάλαιο 3 και 4. Εκεί ε, είναι αυτά τα σημεία. Τα μέτρα τα οποία ε, δημιουργούν πρόβλημα εμπιστευτικότητας απορρίτου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν Ελπίζονται λαμβάνοντας υπόψη αρχή της αναλογικότητας και τους περιορισμούς. Θα πρέπει η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο των επικοινωνιών να είναι εγγυημένο. Έτσι θα υπάρξει εμπιστοσύνη από πλευρά καταναλωτών. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση για να μπορέσουμε ε, σε αυτή τη συνδεδεμένη ήπειρο να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Στρέφομαι στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Madam, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τον εισηγητή ότι το απόρριτο των επικοινωνιών και προστασία του ιδιωτικού βίου καθώς και των προσωπικών δεδομένων είναι καθοριστική σημασία για να υπάρξει εμπιστοσύνη από την πλευρά των καταναλωτών και αξιοπιστία στην ενιαία αγορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω έχει δώσει, αποδώσει τη προσοχή στα θέματα αυτά στην πρότασή της. Νομίζω λοιπόν ότι λίγο πολύ ακολουθούμε το σκεπτικό του εισηγητή. Ίσως λίγα σχόλια τεχνικού χαρακτήρα για τις τροπολογίες που είδαμε να περιλαμβάνει η έκθεση. Κατά πρώτον, φαίνεται να υπάρχει παρανόηση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τι χρειάζεται να διαχειριστής της κυκλοφορίας, ελεγκτής της κυκλοφορίας. Όταν διαβάσει κανεί τι τροπολογίε, καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και στον έλεγχο τη κυκλοφορία οι ίδιε αρχέ εποπτεία που ούτω ή άλλω ισχύουν. Αλλού όμω δεν ισχύει αυτό. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αναφέρει ρητό Συγκεκριμένε τεχνικέ επιθεώρησης, διότι θέλουμε να είμαστε τεχνολογικώ ουδέτεροι στην πρόταση. Να ισχύουν οι βασικές αρχές. Υπ' αυτήν είναι λοιπόν κάποιε τοπολογίε, παρόλο που επιδιώκουν τον κοινό στόχο που έχουμε μαζί σας, ίσως είναι κάπως εσφαλμένα διατυπωμένε, κάπω παραπλανητικά. ένα άλλο επίση γενικό ίσω σχόλιο, η αναφορά που έκανε ο την σχετική νομοθεσία για τον ιδιωτικό βίο για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουμε αντίρρηση ω προς την αναφορά αυτή ή καθεαυτή. Απλώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναθεώρηση η σχετική νομοθεσία. Ίσως λοιπόν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον να, κάνουμε λίγο, να κάνατε λίγο για παρατηρήσεις ή σχόλια ώστε να μην υπάρχουν αλλαγές που εντωμεταξύ καταστήσουν το κείμενο αντιφατικό με τα όσα θα ισχύουν. Ευχαριστούμε κύριε Τράβα. Στρέφομαι και πάλι προς τον εισηγητή. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να σχολιάσω το ζήτημα της ε, παρακολούθησης, της εποπτείας. Έχουμε επαφέ με διαφορετικές ομάδες και έχουμε πολλούς συνομιλητές και πολλοί έχουν ανησυχίε και νομίζω ότι κατά τη σύνταξη των τροπολογιών μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή για να βελτιώσουμε την διατύπωση των τροπολογιών, ώστε να είναι κατανοητέ. Ιδίω όπω το θέμα τη προστασία δεδομένων. Εκεί που ανησυχούμε για τι διαδικασίε και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων και το περιεχόμενο αυτή, τη δέσμη μέτρων, το τι συζητά δηλαδή το Κοινοβούλιο για να περιλάβει στις γενικές διατάξεις του πακέτου προστασίας δεδομένων, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Θα βρούμε μια κοινή θέση για να την αποστείλουμε στην Επιτροπή Ήτρε και να συζητηθεί και εκεί. Uh, uh, Πρόθεσμια τροπολογιών 16 Ιανουαρίου στις 6 ώρα το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 10 Φεβρουαρίου. Αν θέλει ο Θεός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την επόμενη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ να είστε όλοι παρόντες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Και σας εύχομαι καλό απόγευμα και κύριε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασεβούργο.